και περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη που είναι η έκθεση τη κυρία Φωτίγκα. Συνέχεια που έχει δώσει η ΕΕ στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση τη προπαγάνδα εναντίον τη από τρίτου. Κύριε Σιγητέ, κύριε Φωτίγκα, έχετε τέσσερα λεπτά. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, έχω την τιμή να παρουσιάζω τις συστάσεις προς το Συμβούλιο και την ύπατη εκπρόσωπο για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Τέσσερα χρόνια μετά από την υιοθέτηση, την έγκριση της μαρικής έκθεσης για την Stratcom της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αντιμετώπιση δηλαδή της εχθρικής προπαγάνδας κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τρίτα μέρη. Ήμουν εισηγήτρια για την άλλη έκθεση επίσης Θέλω να υπενθυμίσω ότι η πρώτη έκθεση εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2016. Είχε δύο μέρη που αναφέρονταν στους βασικούς πρωταγωνιστές, στους βασικούς παίκτες αν θέλετε, στην προσπάθεια αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει την εχθρική προπαγάνδα από τρίτα μέρη. Πρόκειται για κράτη, την Ρωσική Ομοσπονδία κατά κύριο λόγο, αλλά και για μη κρατικού φορείς κυρίως ε, ριζοσπαστικοποιημένους φορείς όπως ο ISIS. Αυτή τη φορά οργανώσαμε λίγο καλύτερα τις συστάσεις μας με τρόπο εν τέλει διαφορετικό χάρη στις συνεισφορές από διάφορες πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι, διαχωρίσαμε την έκθεση πρώτον στην κατάσταση το 18 Αναφερόμαστε στον ευρύδικο πόλεμο που αντιμετωπίζουμε. Τονίζουμε εν συνεχεία την αναγκαιότητα να αποφύγουμε τη λογοκρισία στην προσπάθεια αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των ψευδοειδήσεων. Αυτές τις στάσεις που βάλουμε στα κράτη-μέλη και στο Συμβούλιο. Τονίζουμε την αναγκαιότητα ποιοτική δημοσιογραφίας, την σημασία της ελευθερίας του λόγου και των μέσων. Επίσης, τονίζουμε την δυνατότητα λήψης νομοθετικών μέτρων ή κανονιστικών μέτρων σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ακόμα και στο ανθρωπιστικό δίκαιο θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τον πόλεμο στον κυβερνοχώρο ή τον πόλεμο στο επίπεδο των πληροφοριών. Τονίζουμε επίσης την διαφοροποιούμενη κατάσταση όσον αφορά τους πρωταγωνιστές αυτού του παιχνιδιού, το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης ορισμένων ε, φορέων και μερών, την εμφάνιση δημοφιλών ιστοτόπων που προάγουν την ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας, την διάδοση των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, που είναι και αυτά ιδιαίτερα δημοφιλή. Πολλά λοιπόν έγιναν από τότε στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε διάφορους άλλους φορείς αλλά και στην κοινωνία των πολιτών τα τελευταία δύο χρόνια. Στην έκθεση επίσης αναφέρουμε αυτές τις δραστηριότητες και τονίζω προκειμένου της, ε, τη σημασία της αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης τη σημασία αυτών των πρωτοβουλίων για τη δημοκρατία καθώς και τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας και της συνεργασίας με ομοειδάτες χώρες. Στο δεύτερο τμήμα αυτής της έκθεσης διαλαμβανόμεθα των διαφόρων τύπων παραπληροφόρησης και εχθρικής προπαγάνδας και στο τρίτο μέρος μιλούμε για την προστασία των επικειμένων εκλογών μας, των ευρωπαϊκών εκλογών, των εκλογών του 2019. Το 2019 είναι έτος 29 διαφορετικών εκλογών σε διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται οι ευρωπαϊκές εκλογές βεβαίως που θα γίνουν ταυτόχρονα σε ορισμένες χώρες. Ζήσαμε την προσπάθεια παρίσφρησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε διάφορες εκλογές και δημοψηφίσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και αλλού. Πρέπει λοιπόν να αποδειχθούμε ανθεκτικοί εναντί αυτών των προσπαθειών εμπλοκής Ο ρόλος της Stratcom East λοιπόν προκειμένου θα είναι πολύ σημαντικός. Και αναφέρουμε και σε δύο άλλες task force. Αναφέρουμε σε αυτήν για τα Δυτικά Βαλκάνια και σε αυτήν για την ε, Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο Κύριος Μίμητσακ, μέρος της Αντιπρόεδρου της Κομισιόν, είπα της εκπροσώπου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτέ, σας ευχαριστώ πολύ που διαθέσατε χρόνο για να συζητήσετε ε, αυτά τα ζητήματα παραπληροφόρηση ε, και ξένη παρέμβαση. Πάρα πολύ επίκαιρα θέματα εν ώψη των ευρωεκλογών. Σα ευχαριστώ όλου ε, για την συνεισφορά σα και ιδίω θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Νίλ Σπιέτα Φωτίγκα που τόσο επίκαιρα κάνει αυτέ τι τόσο εύστοχε συστάσει που συμβαδίζουν με τη λογική και τι δράσει του σχεδίου δράση κατά τη παραπληροφόρηση που υπέβαλε, είπατε, εκπρόσωπος ε, ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η ανταπόκρισή μας ε, και η αντίδρασή μας σε αυτές τις κυβερνοαπειλές είναι κοινή δράση. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις προσπάθειές μας, αλλά θα πρέπει και τα κράτη-μέλη συλλογικά να αναβαθμίσουν τις προσπάθειές τους, όπως λέει στα συμπεράσματά του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ε, στις συστάσεις γίνεται λόγος για το πόσο κομβική σημασία έχει η ελευθερία έκφρασης, ελευθερία λόγου, ο πλουραλισμός ε, για τις ανθεκτικές ε, κοινωνίες διότι οι θεμελιώδεις αξίες μας πραγματικά πρέπει να είναι ε, στο επίκεντρο ε, της μάχης που θα δώσουμε κατά της παραπληροφόρησης. Αυτό είναι ακριβώς το πνεύμα με βάση το οποίο καταρτήσαμε και τώρα εφαρμόζουμε το σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης. Η έκθεση καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εξασφαλίσουν ότι η στρατηγική επικοινωνία της Ένωσης θα λάβει ύψιστη προτεραιότητα και ότι τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη της Ένωσης θα συνεργαστούν στενά για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης αυτής. Και μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω ότι όλα αυτά ήδη συμβαίνουν. Όμως, είναι μια μακρόπνοη προσπάθεια που υπερβαίνει τις ευρωεκλογέ του τρέχοντος έτους. Γι' αυτό και βασιζόμαστε στην συνεχή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από πλευράς δημοσιονομικής. Με το σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης αυξάνουμε τη στελέχωση των τριών ειδικών ομάδων ε, για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, για να μπορούν να ανοιχνεύουν, να αναλύουν και να ε, καταγγέλουν την παραπληροφόρηση, να ευαισθητοποιούν για τον αρνητικό αντίκτυπο, κυρίως όμως ε, να βελτιώνουν τον τρόπο επικοινωνίας και μετάδοσης των αξιών και των πολιτικών μας. Την επόμενη εβδομάδα θα δρομολογηθεί το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, όπως λέει το σχέδιο δράσης, ένα σύστημα που θα καταστήσει πιο εύκολο για τα κράτη-μέλη να ανταλλάσσουν εκτιμήσεις, δεδομένα και βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης εν των ευρωεκλογών. Αυτό θα βελτιώσει ε, την ευαισθητοποίηση, θα προωθήσει κοινέ δράσει, κοινή αντίδραση εφόσον χρειαστεί, ακόμη και σε ό,τι αφορά την αύξηση τη ευαισθητοποίηση και την μεγαλύτερη ανθεκτικότητα τη κοινωνία. Εκτιμώ το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το έργο ε, των ειδικών ομάδων Stratcom και σε ό,τι αφορά ε, την επικοινωνιακή πολιτική και τη μάχη τους κατά της ε, παραπληροφόρησης για τα Δυτικά Βαλκάνια ε, και το Νότο επίσης έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά αυτές οι ειδικέ ομάδες. Η Stratcom έχει καταλογοποιήσει, έχει αυξήσει να αυστοποιήσει για πάνω από 5.000 περιπτώσεις παραπληροφόρησης από ρωσικές πηγές. Δυστυχώς αυτός ο αριθμός ε, θα αυξηθεί κατά πάσα πιθανότητα πολύ περισσότερο. Δεν θα ε, φύγει το πρόβλημα αυτό, δεν θα λυθεί σύντομα από ό,τι φαίνεται. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνουν απαλλαγμένε από ξένε παρεμβάσει οι ευρωεκλογέ και ένα τρόπο να το πετύχουμε αυτό είναι ε, αυξάνοντα την ευαισθητοποίηση για τι προκλήσει ε, που υπάρχουν με στενή συνεργασία με τα μίντια, κοινωνία των πολιτών, πλατφόρμε μέσων κοινωνική δικτύωση μεταξύ άλλων. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση εργάζεται σε πλήρη συντονισμό με το Κοινοβούλιο και τις υπηρεσίες της Κομισιόν. Φυσικά, το σχέδιο δράσης θα σεβαστεί πλήρως τις εθνικές προσεγγίσεις, την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία ε, των μέσων ενημέρωσης που θα καθοδηγούν τις δράσεις μας. Ταυτόχρονα, βελτιώνουμε τη συνεργασία μας για την αντιμετώπιση ξένων παρεμβάσεων και υβριδικών απειλών με τους διεθνούς μας εταίρους όπως είναι το ΝΑΤΟ και η ομάδα των 7, το G7. Συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Ήδη εξελίσσεται. Ανταλλάσσουμε εκθέσει εκτίμησης ε, για το περιβάλλον των πληροφοριών. Ε, συντονισμένες δράσεις αναλαμβάνουμε. Ασκήσεις ε, με σενάρια κάποιων ευρυδικών απειλών. Επίσης, θα πρέπει να συνεργαστούμε ακόμα περισσότερο με τι γείτονε χώρε για να προωθήσουμε το θεματολόγιο τη Ένωση. Θέλουμε να επενδύσουμε στη θετική επικοινωνία, στη δημόσια διπλωματία στι χώρε γειτονία. Αυτό είναι σημαντικό αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση και να προωθήσουμε τι κοινέ αξίε και τα κοινά συμφέροντα. Η δημόσια διπλωματία και η στενή συνεργασία με τι αποστολέ αντιπροσωπή της Ένωση ε, επιτόπου είναι πολύ ισχυρά εργαλεία που προβάλλουν μια θετική εικόνα της Ένωσης στον κόσμο. Το καλύτερο αντίδοτο στην παραπληροφόρηση αφενός είναι ένα υγιές περιβάλλον ε, για τα μέσα ενημέρωσης και αφετέρου η προβολή των ε, θετικών ενωσιακών πολιτικών. Οι πολίτες μας έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση σωστές πληροφορίες, όχι ψευδείς ειδήσει. Έχουν το δικαίωμα σε ένα πλουραλιστικό δημοσιογραφικό περιβάλλον, σε ποιοτικέ πληροφορίες. Γιατί μιλάμε για την ποιότητα της δημοκρατίας μας, για την ποιότητα της Ένωσής μας. Ευχαριστώ. E, e, Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε την κυρία Φωτέγκα για την ε, εξαιρετική της έκθεση. Είναι ένα κείμενο που αναγνωρίζει την ε, σημασία των ε, εκστρατιών προπαγάνδας και της ανάγκες να τις καταπολεμήσουμε. Ιδίω όπου υπάρχει κατασκοπία από τρίτες χώρες. Πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 100 ε, μελών και προσπάθειες σωστής ενημέρωσης. Ο πόλεμο στο επίπεδο τη πληροφόρηση είναι ε, περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Πρέπει να δράσουμε γέρο και να μην ξεχνάμε ότι. Ο Καζίμοφ μίλησε ήδη από το 2013 για την ε, σημασία και το πόσο επίκαιρο είναι, είναι το ψηφιακό επίπεδο στην σε ό,τι τα πολεμικά πράγματα. Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να διαχωρίζουμε σωστά τα ψεύδια από την αλήθεια. Γιατί είναι ένα νέο τρόπο να διεξάγεται πόλεμο. Και μάλιστα έλεγε ο ίδιο ότι υπάρχουν κάποιοι που χρησιμοποιούν όλο το ταλέντο σε αυτό το επίπεδο για να πετύχουν του πολεμικού του σκοπού. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σε φροντιακή συνεννόηση και με τον ΝΑΤΟ και το G7 για όλα αυτά τα θέματα. Το να παραμείνουμε αδρανείς θα σημαίνει απειλή εις βάρος 500 εκατομμυρίων πολιτών και υπονόμευση των αξιών και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε και τώρα ε, ε, τους σοσιαλιστές και δημοκράτες ο κύριος Φρόιντ. Ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο παραπάνω από δύο μήνες ε, γίνονται εκλογές στην Ευρώπη και όπως και με το Brexit, με την εκλογή του Αμερικανικού, Αμερικανού Προέδρου ή την εκλογή του Γάλλου Προέδρου, ε, υπάρχουν προκλήσεις και σε αυτή την περίπτωση και σίγουρα στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ε, υπάρχει το πρόβλημα της παραπληροφόρησης, ε, προπαγάνδας και των ψευδών αυτών ειδήσεων που θα κατακλείσουν, που θα μεταφέρουν πληροφορίες προπαγάνδας και θα είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε ξεχωρίσει κανείς το ψέμα από την αλήθεια ε, την πληροφορία από την ε, προπαγάνδα και νομίζω ότι πραγματικά είναι σημαντικό που ασχολείται με την αντιμετώπιση παραπληροφόρηση και των ψευδών ειδήσεων η ΕΕΔ. Αυτό όμως είναι ένα πρώτο βήμα. Το πρόβλημα εγώ που βλέπω είναι ότι η τεχνολογική ε, πρόοδος μας έχει ξεπεράσει κατά πολύ όπως και συνεχίζει να κάνει. Ε, εμείς ε, προσπαθούμε να παλέψουμε με προχθεσινά μέσα και όπλα τη χθεσινή παραπληροφόρηση, ενώ η προπαγάνδα έχει προχωρήσει πιο πέρα. Πρέπει λοιπόν ε, να δούμε τι είναι ήδη στην αγορά και πώς θα είναι το μέλλον και υπάρχουν ε, δυσκολίες κανείς ε, να διακρίνει ένα βίντεο αν είναι ε, κατασκευασμένο, αν είναι πραγματικό ε, και αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τώρα την έκθεση θέλω να ευχαριστήσω όλους τους και που συνεργάστηκαν για την εκπονησή της. Είναι η τελευταία φορά που βρίσκομαι εγώ εκπρόσωπος της Αυστρίας Βρήκα πολύ αυτά τα πέντε χρόνια ε, και θα ήθελα ε, να μην ε, επηρεαστεί και να μην φρεναριστεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση από εθνικιστικές ή αντιευρωπαϊστικές τάσεις. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, εκ μέρους της ΕΣΥΑΡ, κύριος Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, συγχαρητήρια στην κυρία Φορτάκα για την εξαιρετική έκθεση. Εμείς είμαστε οι φυλακή, ξέρετε, όσον αφορά το θέμα. Και όταν είσαι μπροστά, έτσι είναι τα πράγματα. Έχεις έναν χώρο, ο οποίος είναι επιδεκτικός εκμετάλλευσης από όσους δίνουν τη μάχη κατά της ελευθερίας υποκινούμενοι πολλές φορές από τρίτες χώρες που δεν αξίζει καν να αναφέρω. Στην πολιτική ζωή έχουμε όμως ευκαιρία να κάνουμε κάτι. Έχουμε εκλογές. Και το Brexit μπορεί να είναι μια ευκαιρία για αλλαγή. Και υπάρχουν και άλλες συγκυρίες οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία για μας. Ξέρουμε βέβαια ότι υπάρχουν ευκαιρίε και για του άλλου. Ευκαιρίε που θα αξιοποιήσουν, θα εκμεταλλευτούν οι εχθροί τη ελευθερία, οι εχθροί τη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Και τώρα, εκ μέρου των φιλελευθέρων, ο κ. Αυστρεβίτσιο. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η πρόσβαση στην πληροφορία είναι όλο και πιο επικίνδυνη, πιο επιδεκτική σε ψευδοειδήσει. Τα κρατημέλικοι κυβερνήσει, συνεχίζουν να αγνοούν ή να αρνούνται την ύπαρξη εχθρική προπαγάνδα. Πρέπει επιτέλου να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα, να αξιολογήσουμε την απειλή στην επικράτεια της Ευρωπαϊκή Ένωση και να λάβουμε μέτρα με τρόπο δραστικό για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ψευδοειδήσεις. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τα ψέματα, την προπαγάνδα, την παραπληροφόρηση, τις ψευδοειδήσεις, όλα αυτά που προέρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν διαφόρων ειδών τρομοκρατίες. Υπάρχει στρατιωτική τρομοκρατία, υπάρχει τρομοκρατία κατά της κοινωνικής συνοχής. Λοιπόν, Όλα αυτά είναι απειλέ κατά τη δημόσια τάξη. είναι απειλέ κατά των αξιών και τη ζωής των δικών μας κοινωνιών. Και όλα αυτά συνδέονται με τον υβριδικό πόλεμο κατά των κοινωνιών μας, κατά της καρδιάς και του μυαλού των πολιτών μας. Δίνουμε λοιπόν μια μάχη. Έχουμε μια μάχη μεταξύ εξωτικών, μεταξύ ψευδοειδήσεων, αόρατων εχθρών και το πρώτο βήμα που κάναμε ήταν η Stratcom, η Stratcom για να αντιμετωπίσουμε τις ψευδοειδήσεις. Χρειάζεται να λάβουμε αποφάσεις γρήγορα μέσω αυτής της ομάδας Cruise, ε, η οποία πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με ακόμη περισσότερα κονδύλια. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και τώρα για τους πράσινους η κυρία Ρεμπέκα Χάνος. Κύριε Αξιότιμε, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, οι εκπρόσωποι των ομάδων στις διαπραγματεύσεις ε, της ε, έκθεσης ε, της δεύτερης κύρια ήταν ε, πολύ πιο ε, σύμφωνη σε σχέση μεταξύ του σε σχέση με την επεξεργασία της πρώτης έκθεσης. Τώρα θέλουμε να καταπολεμήσουμε την προπαγάνδα και τη ρητορική μίσους και στις περισσότερες περιπτώσεις η χώρα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η Ρωσία που έχει θύμα όχι μόνο την Ουκρανία αλλά το Κρεμλίνο κάνει όλο και και περισσότερες προσπάθειες με και περισσότερα μέσα ε, να επηρεάσει τους Ευρωπαίους πολίτες κατά των κυβερνήσεών τους με τελευταίο παράδειγμα τις διαμαρτυρίες ε, των κίτρινων γυλαίκων κατά των μεταναστών. Ε, υπάρχει λοιπόν παρότρινση μίσους και επίσης επηρεασμός της κοινή γνώμης και για το Brexit μεταξύ άλλων. Όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε γιατί κατά την άποψή μου θα πρέπει να ε, οργανωθεί πολύ περισσότερο η πληροφόρηση, ε, η σωστή πληροφόρηση, να δοθούν ε, περισσότερα χρήματα και οι υπηρεσίες των κρατών μελών ε, και οι σχετικές αρχές ε, να συνεργάζονται ε, και με το ΝΑΤΟ και με τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι χρειάζονται ανεξάρτητα μίντια. Ο πλουραλισμός στις δημοκρατικές κοινωνίες είναι το α και το ω κατά του μίσους, κατά της προπαγάνδας. Επομένως, εδώ πρέπει να δώσουμε τη βάση μας. Ευχαριστώ. Κάσο περμού τώρα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν περάσει ήδη δύο χρόνια από την ε, υποβολή αυτής της έκθεσης. Ε, δεν φαίνεται γιατί έχουμε τα ίδια επιχειρήματα, τις ίδιες καταγγελίες ε, ε, που έχουν ε, ξεγυμνωθεί εδώ και δεκαετίες, σχέσεις καλής και και τα λοιπά. Και βλέπουμε ότι υπάρχει η ίδια βούληση τα λάθη των ιστορικών πολιτικών να τα ρίχνουμε σε ξένους παράγοντες. Ενώ το εκλογικό σώμα είναι αυτό το οποίο τιμωρεί τα πλειοψηφικά κόμματα για τις νεφιλελεύθερες πολιτικές τους και το αποκορύφουμε ότι περιλαμβάνεται στο Ισλαμικό κράτος μια αναφορά που το μόνο που κάνει είναι να χειροτερεύει τις ε, σχέσεις μας με την Ρωσία. Ε, γιατί τη συγκρίνει ουσιαστικά με μια τρομοκρατική ομάδα που καταδικάζει ο, ο ΙΕ. Μιλάμε για δίωξη των δημοσιογράφων. Ε. Μιλάμε για ανεξάρτητη δημοσιογραφία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα είναι ανεξάρτητη. Βλέπουμε ότι η Ένωση ε, ασκεί μόνο κριτική, αλλά ε, δεν ασκεί καμία κριτική σε αυτά που ίδια κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος ευχαριστώ. Συνάδελφοι, είναι αναντήρητο ότι οι υβριδικές απειλές, κυρίως στον τομέα της πληροφόρησης, αποκτούν στρατηγική σημασία για τις κοινωνίες μας. Ιδίως τώρα που τα νέα τεχνολογικά μέσα έχουν αναπτύξει την ε, ταχύτητα και την ένταση των επιθέσεων σε διεθνές επίπεδο με την ε, ε, αλληλοδιασύνδεση που προκύπτει. Όμως, συνάδελφοι, θα πρέπει να κοιτάξουμε, να προστατεύσουμε από τις ψευδείς ειδήσει τους πολίτες, αλλά να μην τους αφήσουμε πεθυμένους σε τρίτους ε, τρομοκράτες ή κράτη ε, στην όλη προσπάθεια μας. Θα, προσπαθήσουμε, θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και την παραπληροφόρηση αλλά και τις απειλές του τζιχάντο ε, online με τον ίδιο τρόπο, με τους κανόνες μας. Θα πρέπει στον τομέα αυτό να μην παραμείνουμε στα τόσα λίγα που έχουν γίνει, ιδίω από τα κράτη που χρησιμοποιούν μέσα πολέμου, πρόξι όπως λέγονται. Θα πρέπει λοιπόν να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στη γεωγραφική διάσταση, γιατί κάποιες φορές είναι ασαφής η ορολογία που χρησιμοποιείται και μερικές φορές μάλιστα είναι και στα όρια της ε, λογοκρισίας. Θα πρέπει λοιπόν να επιβάλλονται κυρώσεις ε, αμερόληπτες και αποτελεσματικές. Ιδάλλως δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σοφοζέρ για την ε, Ευρώπη των Εθνών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Φωτίγκα, δεν ασχολείστε με τη στρατηγική επικοινωνία στην πραγματικότητα. Προτείνετε μέτρα κατασταλτικά για να καταπολεμήσετε μια σαφή προπαγάνδα η οποία προέρχεται από δίθεν εχθρικέ χώρε προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σα εμπνέει η ίδια λογική τη συνωμοσιολογία και των Μπολσεβίκων, τη απειλή των Μπολσεβίκων, όπω τη κυρία Καλνιέτε. Ε, εδώ οποιαδήποτε αντίρρηση στο φιλευρωπαϊκό εγχείρημα το βλέπετε ως προπαγάνδα. Ε, ε, τα κίτρινα γυλαίκα είναι ε, πίσω του η Μόσχα. Το Brexit το Πούτιν. Βρέχει στην Βαρσοβία φταίει ο Πούτιν. Εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε με το κεμαλακισμό που κατακλείζει την Ευρώπη. Φαίνεται να έχετε σταλινιστικές αιμονές. Πότε θα ξαναρθούν τα στρατόπεδα συγκέντρωση. Εδώ λέτε ότι είναι προδότες όσοι δεν συμφωνούν με αυτές τις ιδέες. Προδοσία είναι να ε, θέλουμε να εργαστούμε για μια Ευρώπη χριστιανική που θα συνεργαστεί και με τη Ρωσία για να τη δημιουργήσει. Που θα εμπνέεται για έναν κόσμο ο οποίος θα λειτουργεί ε, χωρίς καμία ψυχή. Τι θέλετε, η Ευρώπη να μην έχει ψυχή ούτε ρωσική ούτε καμία. Ευχαριστούμε. Ο κύριος... Έχετε λάβει γαλάζια κάρτα. Από τον κύριο Τάραντ. Τη δέχεστε. Κύριε Τάραντ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Σοφοζέρ, συμφωνείτε μαζί μου ότι το να συγκρίνετε την κυρία Καρνιέτε με το σταλινισμό και όλα τα άλλα που είπατε είναι κάπως ε, μη αρμόζων διότι όπως εγώ γνωρίζω γεννήθηκε σε σιβηρικό γκούλαγκ. Είναι μια πλήρω, απαντήστε. Παρακαλώ. Ε, κοιτάξτε, ε, χθε ε, συζήτησα με την κυρία Καλνιέτε και γνωρίζω για τις εμπειρίες της από τον Κούλακ. Δυστυχώς δεν μ' άκουγε ενώ μιλούσα. Και της είπα ότι ως προς τη Ρωσία θα πρέπει να παρέμβουμε όχι μόνο λόγω συγκινησιακών ε, καταλήπων ή από ε, εκδικητικότητα, αλλά αναλύοντας ψυχρά και αντικειμενικά την κατάσταση. Και μπορώ να πω ότι και εγώ πολέμησα κατά του κομμουνισμού και ότι το 89 εδώ στο Στρασβούργο συγκεντρώσαμε όλες τις αντικομμουνιστικές δυνάμεις πριν την πτώση του τείχους. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε Σοφοζέρ, αλλά Πρέπει να συνεχίσουμε την ε, διεξαγωγή τη συζήτησή μα κανονικά. Ο λόγο στον κύριο Φουντούλη για ένα λεπτό. Α πούμε μια φορά την αλήθεια μέσα σε αυτή την αίθουσα. Δεν σα ενοχλεί η προπαγάνδα, κύριε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Άλλωστε, από την ίδια την Ένωση εκπορεύεται το μεγαλύτερο ποσοστό προπαγάνδα που κατευθύνεται προ του πολίτε. Σα ενοχλεί μόνο οτιδήποτε στρέφεται εναντίον των δικών σα συμφερόντων. Η Ένωση χρηματοδοτεί εκατοντάδε μη κυβερνητικέ οργανώσει, οι οποίε προπαγανδίζουν τα ιδεολογήματα των κρατούντων αυτή τη στιγμή σχηματισμών μάλιστα είχατε το θράσος να βαφτίσετε τις δικές σας πεποιθήσεις ως αξίες της ενώσεως χωρίς ποτέ βέβαια να ερωτηθούν οι πολίτες των κρατών μελών για κάτι τέτοιο. το χειρότερο όμως είναι πως με τη στάση σας αυτή αποδεικνύεται το γεγονός πως θεωρείτε τους πολίτες ανίκανους να κρίνουν τις πληροφορίες που δέχονται και να επιλέξουν τις θέσεις που τους εκπροσωπούν. αντίθετα με μια πατερναλιστική λογική θεωρείτε πως μόνο εσείς μπορείτε να τους υποδείξετε τη σωστή εντός εισαγωγικών άποψη για εσά οι πολίτε είναι ελεύθεροι να ψηφίζουν ό,τι θέλουν αρκεί να συμφωνεί με εσά. για εμά οι πολίτε τη ένωση έχουν το νου και τη γνώση να κρίνουν και να αποφασίζουν ποιο του αντιπροσωπεύει. ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Καλνιέται για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εάν υπάρχει μία σύσταση που θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά, θα ήταν κατεπηγόντως η ομάδα δράσης για τα θέματα της Ανατολικής Δονίας να γίνει μια διαρκής, ε, ένα όργανο που να λειτουργεί διαρκώς με την απαραίτητη χρηματοδότηση και το απαραίτητο προσωπικό, την απαραίτητη επάνδρωση, στελέχωση. Θα πρέπει επίση να συνεχίσουμε να στηρίζουμε το την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση για τη Δημοκρατία. Ε, το καταπίστευμα δηλαδή, για να υπάρξουν ανεξάρτητα ρωσικά μέσα ενημέρωση. Ε, και ε, αυτό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτό. Θα πρέπει όλα τα πολιτικά κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίση να είναι ω προ τι δωρεές που δέχονται. Θα πρέπει να ξέρουμε ποια κόμματα απευθεία ή εμέσως ε, ε, χρηματοδοτούνται από τι ρωσικέ μυστικέ υπηρεσίε ή τι μεγάλε εταιρείε τη Ρωσία, του μεγάλου ομίλου, για να γίνουν τα παραθυράκια από που θα μπορούν να προωθήσουν τα όχι και τόσο δημοκρατικά του συμφέροντα εκείνοι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα η κυρία Γουόρντ για ένα λεπτό. Η προπαγάνδα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι απλώς για ακροδεξιούς ευρωσκεπτικιστές που έχουν ε, γεννηθεί και τραφεί εδώ και θέλουν να καταστρέψουν το όνειρο ειρήνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανακάλυψε όταν εργάστηκε για την έκθεση το 2016 για το θέμα αυτό, έχει να κάνει με τη Ρωσία και τις χώρες που δεν συμμερίζονται στις ευρωπαϊκές αξίες αυτό το θέμα. Ε, επηρεάστηκε το ε, ψήφισμα το 2016 από τις υπηρεσίες του Πούτιν και αυτές του μπορεί να έχουν τεράστιο αντίκτυπο και στι επερχόμενε ευρωεκλογέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να λάβει μέτρα αυστηρά. Θα πρέπει να ε, ε, υπάρξουν περισσότερα εργαλεία από τι τεχνολογικέ εταιρείε για τον εμπλουτισμό τη προπαγάνδα και να γνωρίζουμε κατά την ταυτότητα όσων χρησιμοποιούν τι πλατφόρμε. Να σβήνονται τα σχόλια που ε, δεν ξέρουμε τι οικονομικά συμφέροντα τα στηρίζουν. Επίση, χρειαζόμαστε περισσότερη ευαισθητοποίηση σε πολιτικό επίπεδο. Λόγω χάρη, ο κύριο Γάλλο ακροδεξιό βουλευτή, έκανε δώρα στην κόρη του Πούτιν και στον εκπροσωπό του εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτά θα πρέπει να απαγορεύονται. Επίση, ε, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αγνοεί την εχθρική προπαγάνδα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια τη προεκλογική εξετρία για τον Brexit. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε τα ε, χρήματα από την παραοικονομία και όλα αυτά που χρηματοδότησαν αυτή την εκστρατεία. Σα ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ να παραμένετε στο χρόνο μιλία σα και τώρα για ένα λεπτό ο κύριο Κρίστιαν Πρέντα. Ευχαριστώ. Η αντιμετώπιση της προπαγάνδας ε, προαπαιτεί το να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς της προπαγάνδας. Και διαφέρουν αυτοί από τη μια χώρα στην άλλη. Στη Ρουμανία, λόγω χάρη, ένας πρώην σοσιαλιστής πρωθυπουργός διαδίδει ψεύδι υποστηριζόμενος από έναν αξιωματικό του κοκκινού στρατού, πρώην αξιωματικό του κοκκινού στρατού. Ε, η κυβέρνηση λοιπόν να διαδίδει ψεύδι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο ο μηχανισμός επαλήθευσης των ε, ειδήσεων χρέωσε το Υπουργείο να πάρει θέση και να πει ε, εντάξει πρόκειται για ε, νοθευμένες ειδήσει τελικά. Ε, κακικό έλεγχο των ε, πηγών. Η κυρία που η Πρωθυπουργός, είναι στη Σπούτνικ κάθε εβδομάδα. Πολλοί πολιτικοί έχουν καταδικαστεί για διαφθορά και υπάρχει... Ε, γίνεται κουβέντα για το πώς απειλεί το κάτω δικαίου της χώρας ο Τζόρτ Σόρος και πώς επίσης είναι κακό πράγμα η δημοκρατία στη Ρουμανία. Αυτό αρχίζει να κατακλείζει την κοινή γνώμη. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο κάθε χώρα όπως και στη δική μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ο μιλητής ο κ. Πιτσούλα για να λεπτό. Cambridge Analytica, Το σκάνδαλο της Cambridge Analytica απλώς επιβεβαιώνει πώς ε, μπορούν να επηρεαστούν εκλογές και δημοψηφίσματα. Αναμένουμε βεβαίως περισσότερη ενημέρωση από το Λονδίνο, να δούμε πραγματικά ε, τι συνέβη και με το Brexit. Δεν μπορούμε λοιπόν να υποτιμήσουμε την εμπλοκή της παρεμβάσεις των Ρώσων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν πρέπει λοιπόν να υποτιμούμε την απειλή. Ίσα ίσα πρέπει να δούμε τι γίνεται στα Βαλκάνια, τι γίνεται με τις υποψήφιες χώρες. Φυσικά δεν είναι μόνο η Ρωσία. Οι ψευδοειδήσεις προέρχονται και από δυτικέ πηγές αλλά και από αλλού. Ο στόχος τους όμως είναι ένας, να καταλύσουν τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνουμε τώρα λίγο πριν από τις εκλογές να δώσουμε αληθή πληροφορία στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το υπαριθμό 1. Ευχαριστώ. Κύριε Σκόβατσεφ. Κύριε Πρόεδρε, λέει κύριο Σκόβατσεφ. Αντιμετωπίζουμε όντως υβριδικό πόλεμο. Πρέπει να λάβουμε μέτρα. Τα εφιστάμενα μέτρα δεν είναι επαρκή. Η East Stratcom η ομάδα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, να γίνει μια ανεξάρτητη ενισχυμένη διεύθυνση με παρκή χρηματοδότηση. Στη Βουλγαρία έχουμε μια τέτοια υπηρεσία υπό την Μαρία Γκάμπριελ. Η βουλιαρκή κυβέρνηση πρότεινε τη δημιουργία μιας τέτοιας υπηρεσίας η οποία θα ενισχύει την ερευνητική δημοκρατία και η οποία θα πατάσει την παραπληροφόρηση και η οποία γενικότερα θα ενισχύει όλους τους φορείς που διεξάγουν πόλεμο κατά των ψευδοειδήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μείνει στο απειρόβλητο πρέπει να καταλάβει πού υστερεί σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστούμε. Κύριο Γκάλερ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στον συνόλεφο Όντιεν Φρόιντ. Συμφωνώ απόλυτα με το 100% των όσων είπε. Αυτό θα του έλεγαν ήταν εδώ, δεν είναι εδώ. Βέβαια, δεν κατάφερε μέσα σε δύο λεπτά να πει ούτε μια φορά τη λέξη Ρουσία. Ρωσία. Δεν ξέρω, ίσως να είναι αυστριακή ιδιαιτερότητα. Τέλο πάντων, τα πράγματα όμως πρέπει να τα λέμε με το όνομά του. Ε, η Ρωσία το μόνο που θέλει να καταφέρει είναι η αποσταθεροποίηση της Ευρώπης, ε, να αποδυναμώσει το mainstream. Όλα τα άλλα είναι ελκυστικά. Οι ΚΕΙ που τότε ΣΕΣΕΔΟΥ ή τώρα Ρωσία είχε τη δική της ιδεολογία έχουν περάσει και η ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας πρέπει να ενισχυθεί. Εκεί που πέφτει το χρήμα, ε, κύριε ε, Σαφάζερ, ε, πρέπει να υπάρξουν νόμοι για να μην επιτρέπεται η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα. Μπορεί να παίξει ένα συντονιστικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και η ομάδα ειδική είστε πρέπει να ενισχυθεί και να υπάρχουν και οι απαραίτητες επαφές και διαδικασίες δικτύωση με εθνικούς συνδέσμους από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον κύριο Ρανζέλ που είναι ο εμόδιο επόμενο ομιλητή. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον επόμενο τον κύριο Κούκαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σοβαρή απειλή στη κατά τη Δημοκρατία. Πώ θα αντιδράσουμε αποτελεσματικά κατά τη προπαγάνδας, παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων από τρίτε χώρε, Όλο και πιο δύσκολα μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό Πρέπει λοιπόν και σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο να προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε τις αξίες μας και να αντιμετωπίσουμε τον κυβερνοπόλεμο και τον υβριδικό πόλεμο. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι ε, όμορες χώρες προς Ανατολάς και προς Δυσμάς και προς Νότον. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε στο περιφερειακό επίπεδο, να βελτιώσουμε την επικοινωνία πάνω στα θέματα που από τον Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητώ επίσης ε, μεγαλύτερη χρηματοδότηση, περισσότερη στελέχωση, περισσότερα μέσα ε, και περισσότερη συνεργασία ε, με τις επίσημους χώρες όπως είναι η αντιπροσωπή της Ένωσης στις τρίτες χώρες. Η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, της εχθρικής προπαγάνδας πρέπει να είναι προτεραιότητα, όχι μόνο για τι ευρωεκλογέ αλλά και ε, εν ώψη και το επερχόμενου Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιόν. Πρέπει καλύτερα να μεταδώσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αλλιώς οι δημοκρατίες μας μπορεί να μην ανθέξουν, να μην επιβιώσουν απέναντι στις εξωτερικές αυτές απειλές και πιέσεις. Ευχαριστώ. Κύριος Κέλα, είναι επόμενο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, το Stratcom έχει δώσει καταπληκτικά αποτελέσματα ε, με 5.000 παραδείγματα να λέει στατιστικά το τι συμβαίνει. Αυτή η ομάδα δράσης λοιπόν του Stratcom θα πρέπει να γίνει μόνιμη ομάδα με τις δικές της, με δικά της κονδύλια και το δικό της προσωπικό. Εδώ λοιπόν ε, θα πρέπει να ε, δώσουμε το πλήρες νόημά του στο στράτικο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια σημαντική αρμοδιότητα για να βελτιώσει τις δεξιότητες και να δώσει τη δυνατότητα απόκρισης ε, στα κρατη και τα θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνεργασία με τον ιδιωτικό κλάδο, να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη και να προωθήσουμε την εκπαίδευση κατά της παραπληροφόρησης θα πρέπει να δώσουμε κατά απαραίτητα κονδύλια στο Stratcom. Θα πρέπει να αναλάβει αυτή την αρμοδιότητα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συντονίσει τις σχετικές προσπάθειες με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Σας ευχαριστούμε ο κύριος Στέτινα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Εδώ έχουμε 38 συστάσεις την έκθεση. Ο στόχος όμως όλων είναι να αντιμετωπίσουμε την προπαγάνδα κρατών. Στο 8, στο προήμιο επίσης, αναφέρονται κύριες πηγές παραπληροφόρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2014 ο Ρώσος στρατηγός Γκερασίμοφ θέσπισε νέες μορφές πολέμου στον κυβερνοχώρο λέγοντας ότι αν επιλέξουμε σωστά τις λέξεις και τις διαδώσουμε με το σωστό τρόπο, ο πόλεμος αυτός θα έχει πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα από τις βόμβες και τις ρουκέτες. Λοιπόν, ας ξυπνήσουμε επιτέλους και ας συνειδητοποιήσουμε ότι χάνουμε τον κυβερνοπόλεμο με τη Ρωσία. Ας πούμε επιτέλους τη, τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Αλλιώς θα χάσουμε σύντομα τις δυνατότητές μας σε αυτόν τον χώρο. Ευχαριστώ. Ε, δεν βλέπω. Ε, κυρία Αντρική Όχι, δεν είναι εδώ. Σουίτσα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Με απασχολεί το θέμα των ψευτοειδήσεων και της παραπληροφόρησης. Ακούμε τόσο πολλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τελευταία κυρίως για τον ρόλο τρίτων χωρών. Λοιπόν, εγώ ανησυχώ και πρέπει όλοι να ανησυχούμε για την κατάσταση. Γι' αυτό είμαι υπέρ της έκθεσης. Θα υπερψηφίσω γιατί διαλαμβάνεται των δυνατοτήτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση και τις ψευδοειδήσεις. Μπορούμε να κάνουμε πολλά σε εθνικό επίπεδο, όμως το διαδίκτυο είναι παγκόσμιο. εννοείται ότι συμβαίνει, συμβαίνει παντού, πέραν των σύνορων. Η προπαγάνδα από την Ανατολή είναι επίφοβη, σίγουρα επηρέασε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στον Εμερ Βασίλειο, τα αποτελέσματα του οποίου φυστάμεθα σήμερα. Όχι μόνο εμεί, αλλά και οι Βρετανοί πολίτε. Ό,τι και να λέμε. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν να πατάξουμε την προπαγάνδα από τρίτους φορείς, από τρίτες ε, χώρες, ιδιαίτερα εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών. Ευχαριστώ. Ζροεύσκη. Πρόεδρε. Στην αρχή της θητείας μας είχα πει δύο λόγια για τον ευρυδικό πόλεμο. Είχα πει ότι ευρυδικός πόλεμος σημαίνει ευρυδική εμπλοκή, ευρυδικά μέτρα. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε την προπαγάνδα, την παραπληροφόρηση, αλλά να διασφαλίσουμε και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τη σωστή εκπαίδευση και την απαραίτητη συνεργασία. Στρατηγική συνεργασία θα έλεγα. Δυστυχώ είμαι σήμερα απογοητευμένο από τα όσα έχει κάνει, μάλλον δεν έχει κάνει η Κομισιόν, διότι ήδη το 2016 είχαμε ζητήσει από την Κομισιόν να κάνει περισσότερα. Η Φορτέγκα είχε αναλάβει πρωτοβουλίες στην Επιτροπή Άμυνας. Η Κομισιόν θα πρέπει να είναι μπροστά από τους διάφορους παίκτες στον χώρο, στον πόλεμο της παραπληροφόρησης, του πολέμου στον κυβερνοχώρο. Δυστυχώς η Κομισιόν τώρα τρέχει πίσω από τις εξελίξεις και μάλιστα ανταποκρίθηκε με μεγάλη καθυστέρηση σε προβλήματα τα οποία ήταν γνωστά στον δημόσιο χώρο εδώ και χρόνια. Οι περίπου 40 συστάσεις είναι καλές εν πάση περιπτώσει, είναι επίκαιρε. Ας κάνουμε κάτι τώρα, χωρίς καμία καθυστέρηση παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Προσέλκυση προσοχής του Προέδρου. Έχετε το λόγο κύριε Αζάρ. Ρανζέλ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που άργησα κύριε Πρόεδρε, αλλά ε, είχα μια συνάντηση με τον κύριο Μπαρνιέ. Καταλαβαίνετε ότι ήταν σημαντικό αυτό και δεν μπορούσα να είμαι εδώ βέβαια. Θα ήθελα κυρίως να πω το εξή. Το θέμα της προπαγάνδας, όλος ιδιαίτερος της προπαγάνδας που στόχο έχει να εξαπατήσει την κοινή γνώμη και όπως γνωρίζουμε συμβαδίζει με την όλη, πάει εν παραλίλω με τη συζήτηση που κάναμε για τις ψευδεί ειδήσει. έρχεται από συγκεκριμένε χώρες. Και εδώ πρέπει να έχουμε μια πολύ αποφασιστική ε, δράση. Να αναχαιτήσουμε κάθε προσπάθεια, τα στρατηγικά συμφέροντα, τα οποία συνήθως είναι κακοπροαίρετα από τρίτες χώρες να επιβληθούν και να επηρεάσουν τις δικές μας προεκλογικές εκστρατείες, τις συζητήσεις μας και το υποψηφίσματά μας. Γι' αυτό λοιπόν η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή η καταπολέμηση αυτού του είδους των προσπαθειών, είναι πολύ σωστή. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο ευρυδικός πόλεμος δεν είναι κάτι το καινούριο. Ωστόσο, οι εξελίξεις έχουν επιταχυνθεί. Έχουν ε, ανοίξει νέοι διαβλή και ακόμα περισσότερο μέρο του κοινού μπορεί να πέσει θύμα προπαγάνδας, γιατί υπάρχει πρόσβαση πιο εύκολη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιοι προσπαθούν να, να επηρεάσουν τις δημόσιες συζητήσει στην Ευρώπη, τη δημοκρατία, ε, γιατί έχουν περισσότερο χρόνο για να... χώρο για μάλλον για να δράσουν. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πω ότι στηρίζω θερμά τι συστάσει αυτή τη έκθεση και παρόλο που σε μια ανεπτυγμένη δημοκρατία θα πρέπει να είναι σαφέ, δεν είναι. Ε, θα πρέπει να υπάρχει και επικριτική ε, δυνατότητα κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, η κριτική μπορεί να είναι και επικοδομητική, δεν είναι κάθε κριτική ε, εχθροπραξία. Όμω πρέπει να τονίσουμε ότι εδώ και πολύ καιρό δεν ακούμε τι φωνέ των πολιτών. Θα πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσει που να εξυπηρετούν και τα δικά του συμφέροντα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Επιτίδιο. Ε, στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από την αλματώδη εξέλιξη τη τεχνολογία, οι αρχέ και οι μέθοδοι τη προπαγάνδα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν με πολλού και διαφόρου τρόπου, οι κυριότεροι από του οποίου είναι η παραποίηση τη αλήθεια και η διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ε, βασική αρχή για μια δημοκρατική κοινωνία να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ε, εχθρική προπαγάνδα είναι η παρουσίαση της αλήθειας στο κοινό και όχι η δίωξη των πολιτικών αντιπάλων και των δημοσιογράφων οι οποίοι ασκούν ε, κριτική στην κυβέρνηση είτε παρουσιάζουν διάφορα σκάνδαλα. σε εθνικό επίπεδο η ενημέρωση του κοινού η αντικειμενική και αμερόληπτη επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας ενός λειτουργικού συστήματος ραδιοτηλεοράσεως πολλές φορές όμως το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί σωστά. αυτό συμβαίνει στην ελλάδα που η ραδιοτηλεόραση εθνική έχει μεταβληθεί σε όργανο κομματικό του κυβερνώντος κόμματος και μάλιστα φτάνει στο σημείο να μην καλεί στις εκπομπές τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές του κόμματος στο οποίο ανήκω της χρυσής αυγής που είναι η τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας. όπως αντιλαμβάνεσαι με τέτοιες μεθόδους υπάρχει αναξιοπιστία και δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε εχθρική προπαγάνδα. ευχαριστώ. E, Ευχαριστούμε. Ροχόνεν Λέρνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα κοινωνικά μέσα και στα παραδοσιακά μέσα η παραπληροφόρηση είναι εξίσου ε, απειλή κατά της δημοκρατίας. Γι' αυτό οι πληροφορίες και οι ειδήσει που λαμβάνουμε πρέπει να είναι ακριβείς και αληθεί. για να μπορούν και οι άνθρωποι να αποφασίζουν σωστά όταν πρόκειται να ψηφίσουν ε, με περιστατωμένη γνώση και επίγνωση. Θα πρέπει λοιπόν όταν εντοπίζονται οι ψευδείς ειδήσει και παραπληροφόρηση στα κοινωνικά δίκτυα να απαιτείται και να απομακρυνθούν, να σβηστούν θα πρέπει να εντοπίζονται στο δυνατόν γρηγορότερα προτού ε, διαδοθούν ε, ευρέως. Θα πρέπει οι πλατφόρμες στο διαδίκτυο να, να καταστήσουν σαφές ότι και οι κανόνες της διαφήμισης που, τη στηρί, που του στηρίζει θα πρέπει να είναι διαφανείς θα πρέπει να μην μπορούν να μετακινούνται τεράστια ποσά λογαριασμών ε, τόσο γρήγορα και τα τεχνολογικά μέσα αλλάζουν διαρκώς. Είναι πολύ εύκολο να στήσει κανείς ένα ψεύτικο βίντεο και ένα ψεύτικο φιλμάκι και οι ψευδείς ειδήσει πρέπει να καταπολεμηθούν με την ε, σωστή ε, γνώση με τον αλφαβητισμό των μέσων και ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Μαριάς κύριε πρόεδρε συζητούμε εδώ για την παραπληροφόρηση την προπαγάνδα τις ψευδείς ειδήσει αλλά αυτά πρέπει να εφαρμοστούν και εναντίον του ίδιου του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου διότι όπως ξέρετε όλοι το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ανέθεσε σε μια δημοσκοπική εταιρεία να κάνει δημοσκόπηση για τις ευρωεκλογέ η οποία δημοσκοπική εταιρεία αντί να κάνει δημοσκόπηση πήρε τις δημοσκοπήσεις σε εθνικό επίπεδο δημοσκοπήσεις που έγιναν για εθνικές εκλογές και έβγαλε συμπεράσματα για το ποιοι εκλέγονται και ποιοι δεν εκλέγονται από αυτή εδώ την ευρωβουλή πόσοι ευρωβουλευτές από εμά δεν θα εκλεγούν και πόσοι δήθεν θα εκλεγούν. αυτό είναι μαύρη προπαγάνδα παραμονές των ευρωεκλογών είναι fake news είναι καθοδηγημένη προπαγάνδα εναντίον συγκεκριμένων ευρωβουλευτών. αυτό πρέπει να καταγγελθεί και να απαγορευτεί και να σταματήσει αυτή την τακτική το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο διότι είναι έσχος και γι' αυτό πρέπει να τοποθετηθείτε όλοι συνάδελφοι να μην επιτρέπουμε τα fake news ότι ορισμένοι δίθεν από εμά δεν θα εκλεγούν επειδή το λέει μια δημοσκοπική εταιρεία και αυτό έχει αναπαραχθεί σε όλα τα μίντια σε όλη την ευρώπη. είναι ντροπή είναι έσχος. Ευχαριστώ πολύ για το παθιασμένο αυτό σας λόγο και τελευταίο στο Catch Κάρσκι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πολλοί είπαν για την παραπληροφόρηση μέσω παραδοσιακών και νέων μέσων ενημέρωσης παραπληροφόρηση έχουμε και εδώ, στο Ευρωκοινοβούλιο, στο πλαίσιο της συζήτηση. Ένας από τους δράστες είναι ο κύριος Σαφοζέρ, που βρώμησε ε, το στόμα του χρησιμοποιώντας ε, ε, το, βάζοντας στο στόμα του το όνομα του Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου ντροπή και όνειδος και είπε ότι δεν τηρούνταν οι συστάσει ε, και τα όσα είπε και τα κηρύγματα του ε, Ιωάννη Πάρτου Δεύτερου. Αυτό πραγματικά είναι ανήθικο. Ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτούς που λένε αυτά. Και φαντάζομαι θα του τα μεταφέρουν το κύριο Σαφοζέρ αυτά που λέω. Μπορεί να μείνει ε, αυτή η ομιλία ε, ως μία από τις ε, πιο εντυπωσιακές, αλλά είναι αποτέλεσμα, είναι προπαγάνδα και παραπληροφόρηση ουσιαστικά. Να ξαναδώσω το λόγο στον ε, κύριο Νίμιτσα για να ολοκληρωθεί έτσι η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα βουλευτέ. Ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Φωτίνκα και του βουλευτέ ε, για τι παρεμβάσει του. Από αυτή τη συζήτηση, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγω είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία έχουμε ένα κοινό ε, συμφέρον και ενδιαφέρον να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της ε, ξένης παρέμβασης και της παραπληροφόρησης ε, ενώπιον των ε, ευρωεκλογών. Είναι λοιπόν αυτή η συζήτηση και μια ευκαιρία για να προβάλλουμε περισσότερο το θέμα και να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση. Ολοκληρώνοντας, θέλω να επαναλάβω για μια ακόμη φορά τις ευχαριστίες μου για τον ρόλο του Κοινοβουλίου που έχει βάλει προτεραιότητα το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Κυρία Φωτίγκα, για να κλείσουμε. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Εδώ μιλούμε για τον δηλητηριασμό των ψυχών των πολιτών μας. Το καλύτερο παράδειγμα ήταν η κατηγορία της χαρά ε, της και μου της ιδέας. Πούτιν ο ίδιος συνεχίζει τις πολιτικές του Στάλιν και το λέει. Το λέει ο ίδιος χωρίς περιστροφές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους κοιόδης εισηγητές για τις συνεισφορές τους. Όλες εξαιρετικές. Είχαμε ουσιαστικό διάλογο για το θέμα σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Θεωρώ ότι το τελικό αποτέλεσμα, χάρη στη δική σας συνεισφορά, θα βοηθήσει τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν την εχθρική προπαγάνδα. Θα ήθελα ιδιαίτερως να ευχαριστήσω τον κύριο Τάνοκ, ο οποίος με βοήθησε σε πολύ δύσκολες στιγμές όταν εγώ αντιμετώπισα μεταξύ άλλων και κάποια προβλήματα υγείας. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ευχαριστώ, λέει Εδώ κλείνει η συζήτηση επί του θέματος, η ψηφορία αύριο.